2013 την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Πρώτο ο εισηγητής κύριος Πυρίνσκι για τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε κράτος μέλος κάνει την αναλογική εισφορά του στον προϋπολογισμό. Και έτσι προστατεύονται τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Επιτροπή Έλεγχου του Προϋπολογισμού ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση, σχετική έκθεση και κατά τις, όμως κατά τις συζητήσεις πριν την ψηφοφορία εμφανίστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς το ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τον προϋπολογισμό δηλαδή. Συζητήθηκε η περίπτωση προστήμων και κυρώσεων εάν είχαν διαπιστωθεί ατασθαλίες, αλλά υπάρχουν δύο ειδών. Μερικές οφείλονται σε διαφθορά, απάτη ή εγκλήματα και άλλες, που είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, οφείλονται σε απλά λάθη μη γνώση του κανονισμού και επομένως οι κυρώσεις πρέπει να συνδυάζονται με στήριξη των κρατών μελών ώστε να είναι σε θέση να αποφεύγουν την ε, απάτη και να μειώνουν τον αριθμό περιπτώσεων που οφείλονται σε λάθη. Η έκθεση του 2013 είναι ενδεικτική. Επί συνόλου 2,14 δισεκατομμυρίων ανομαλιών η μεγαλύτερη μερίδα οφειλόταν σε λάθη. Οι απάτες αντιπροσώπευαν μόνο 309 εκατομμύρια. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω το λεπτό θέμα που είναι η καθυστέρηση ή και άρση ορισμένων πληρωμών, πάγωμα πληρωμών γιατί ζητούμε από την Κομισιόν να εφαρμόσει αυστηρά συνήθως τέτοια μέτρα. Αλλά είναι μονόπλευρη αυτή η προσέγγιση γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της τα βασικά στοιχεία που αφορούν την πρόληψη που μπορεί να γίνει όπως το πνεύμα και το γράμμα των άρθρων του άρθρου 325 τη ιδρυτικής συνθήκης που τονίζει ακριβώς την πρόληψη για την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Είναι ουσιώδες λοιπόν τα κράτη-μέλη να αναφέρουν περιπτώσεις απατών και άλλου είδους ανομαλιών γιατί μόνο με τέτοιου είδους πληροφόρηση μπορούν να ταυτιστούν τα προβλήματα και να ζητηθούν λύσεις για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Η πληροφόρηση όμως για τέτοιου είδους ανομαλίες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να κατηγορηθούν ή να δακτυλοδειχθούν ορισμένες χώρες. Απλώς να διορθωθούν οι ανομαλίες εάν χρειαστεί να επιβληθούν πρόστιμα κυρώσεις και εάν φανεί ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες περισσότερες από άλλες τότε ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι άλλες χώρες μέλη πρέπει να τις βοηθήσουν να γίνει η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και πληροφόρησης και κατάλληλος συντονισμός και εκπαίδευση. Μόνο έτσι θα υπάρξει σωστή προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης όπως εξάλλου προβλέπουν και οι αρχές της σωστής διαχείρισης και έτσι θα πληρωθούν και οι προσδοκίες των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που με βοήθησαν στη σύνταξη της έκθεσης, δηλαδή την συνάδελφο Γιάννα Ποπόβα, την κυρία Κουντρούτσα από τη Γραμματεία των Σοσιαλιστών και τον την συνάδελφο Καστήλιο από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Και τώρα η Επίτροπος Γεωργίευα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πυρίνσκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να καταπολεμηθεί φυσικά η απάτη, γιατί είναι σημείο κλειδί για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στις εργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέτασα την έκθεσή σας και χαίρομαι γιατί για πολλές από τις συστάσεις σας ήδη έχει υπάρξει θετική συνέχιση. Να καταδείξω ορισμένα από αυτά. Πρώτα απ' όλα για την ε, παρουσίαση εκθέσεων για τις παρατυπίες. Συμφωνούμε με το πόρισμά σας ότι πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ απατών και λαθών. Θα έχουμε μηδενική ανοχή για τις απάτες, αναμφίβολα, αλλά εάν πρόκειται απλώς για λάθη Πρέπει να κάνουμε προληπτικές δράσεις, πρέπει να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και εναρμόνιση για όλες τις κατηγορίες δαπανών. Αυτή την εργασία έχουμε ήδη αναλάβει μέσω μιας νέος συσταθήσης ομάδας επιτρόπων που ασχολούνται με τα κύρια θέματα και, του κύριου τομεί και τους κύριους τομείς δαπανών για την πολιτική συνοχής. Επίσης συμφωνούμε με την έμφαση που αποδίδεται στη δημιουργία προληπτικών μηχανισμών και ε, να κάνουμε και έναν απολογισμό το 2018 για το τι θα έχουμε κάνει μέχρι τότε και για το εάν η νέα δομή των ρυθμίσεων για τα θέματα συνοχής αυξάνει την αποφυγή παρατυπιών. Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά αυτά που λέτε για τις δημόσιες προμήθειες. Αναγνωρίζουμε ότι ακόμη οι διαδικασίες δημοσίων προμηθειών ε, είναι πολλές φορές αντικείμενο απατών και διαφθοράς και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνουμε για να προωθήσουμε τη νέα οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους είναι και για μας όμως μια ευκαιρία ως θεσμικά όργανα της Ένωσης να προωθήσουμε τις σχετικές αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό που είναι υποδιαπραγμάτευση ήδη. Ελπίζουμε να καταλήξει σύντομα αυτή η διαπραγμάτευση. Αναγνωρίζουμε ότι έχει θεμελιώδη σημασία απόλυτα ασυμβίβαση στάση κατά της διαφθοράς και θα ακολουθήσουμε τέτοιες πολιτικές στο δεύτερο πακέτο μέτρων κατά της διαφθοράς που θα υποβληθεί του χρόνου. Για τον οργανισμό Όλαφ, το έχω πει επανειλημμένα, είναι ζωτική σημασίας, συστατικό στοιχείο της πάλης μας κατά της διαφθοράς και της απάτης. Συνεργαζόμεθα με τον Όλαφ για να υπάρχει πολύ καλή επαφή με την Εποπτική Επιτροπή του εγώ προσωπικά έχω συμμετάσχει στις εργασίες αυτής της, συνοπτικής, της Εποπτικής Επιτροπής ούτως ώστε να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον και για τον Όλαφ και για την Εποπτική του Επιτροπή για να λειτουργούν σωστά όλα αυτά είναι απόλυτα διαφανή και όσον αφορά το θέμα των στατιστικών εργαλείων και των πορισμάτων των αναλύσεων που γίνονται με βάση την εφαρμογή τους. Επιπλέον, θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανεξαρτησία αυτής της υποπτικής επιτροπής στα πλαίσια της πολιτικής προσωπικού και διαχείρισης των πόρων επί των οποίων θα κάνουμε ε, πολύ σύντομα προτάσεις. Χαιρετίζουμε διάφορα σημεία της έκθεσης για το γραφείο του Ευρωπαίου Ισαγγελέως, τη σχετική οδηγία και ολόκαρδα λέω σας ευχαριστούμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα την στήριξή σας. Χρειαζόμαστε αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τέτοια που να είναι σε θέση να προσθέσει αξία στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι. Θέλουμε το θεσμικό πλαίσιο να βελτιώσει ουσιοδός ε, τα αποτελέσματα της μάχης μας κατά τη διαφθορά, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Τώρα από πλευρά τη Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Αριμό. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Επίτροπε, επειδή οι δημόσιοι πόροι είναι περιορισμένοι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, πρέπει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να αντιμετωπίζονται σωστά. Κάθε λεπτό που μας δίνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, λεπτό του ευρώ, πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιείται σωστά. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Αυτά που λέγονται για παρατυπίες κάνουν ζημιά στη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν ζημιά γενικότερα στην αξιοπιστία των πολιτικών γενικότερα λοιπόν. Οπότε, στην ουσία δίνουμε επιχειρήματα σε αυτούς που είναι εχθροί της δημοκρατίας και της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό και για τον τομέα μου της συνοχής. Τα διαφροντικά ταμεία πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιούνται σωστά. Γιατί είναι ένας τομέας πολιτικής όπου έχουν σημειωθεί περισσότερες παρατυπίες. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Κατά την περίοδο που εξετάζουμε είχαμε 321 περιπτώσεις παρατυπίας ε, πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και σε άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε δολιότητα είχαμε 400 και παρατυπίες, όλες μαζί οι παρατυπίες και οι απάτες ανέρχονται σε ύψος 1,36 δις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με βάση αντικειμενικά κριτήρια για να αντιμετωπίζονται παντού οι περιπτώσεις απάτης και δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια μέχρι στιγμής. Επίσης, διαπιστώσαμε μια σειρά παρατυπίες οφείλονται στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Άρα χρειάζεται διοικητική απλούστευση. Για την πραγματική όμως απάτη πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια στρατηγική καταπολέμηση της διαφθοράς και των απατών, όπου πρέπει να έχουμε ακριβώς και πάνω απ' όλα εξωτερική έλεγχη και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι ευρωπαϊκές προκηρύξεις. Πολύ συχνά είναι πηγή παρατυπιών, το είπατε κι εσείς η οδηγία για τις ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να μειώσουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό η οδηγία πρέπει να μεταγραφεί στο εθνικό δίκαιο τάχιστα. Μπορούμε να το επιτύχουμε όλες οι αγκληματικές ενέργειες να έχουν λιγότερες δυνατότητες να περάσουν. Όπως είπα και εγώ, κάθε ευρώ πρέπει να αξιοποιείται σωστά. Το οφείλουμε στους ε, φορολογουμένους. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τη γενική συζήτηση από τις πολιτικές ομάδες θα δεχτώ πολιτικές κάρτες. Τώρα να δώσω το λόγο από πλευρά τη Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ στην κυρία Μακοβέη δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Στην έκθεση αυτή φύγεται το σημαντικότατο θέμα της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δηλαδή των χρημάτων μας, του καθενός από εμά του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Δικά μας λεφτά είναι αυτά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων μας, των πολιτών μας που πληρώνουν από την τσέπη τους, από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς για να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός. Και αυτό ισχύει για όλους. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκά δημοσιονομικά συμφέροντα αφηρημένα. Είναι τα χρήματα των πολιτών. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και πού πηγαίνουν τα χρήματα, διότι αν η προστασία αυτών των χρημάτων. Γίνεται σωστά από μια χώρα, όχι τόσο σωστά από άλλη χώρα, τότε υποφέρουν όλοι. Δεν σημαίνει ότι αν σε 10 χώρες μέλη δεν υπάρχουν, δεν σημειώνονται απάτες, όλα είναι εντάξει. Όλοι σημειώνουμε αν υπάρχει απάτη. Και ευχαριστώ την Κομισιόν και την Επίτροπο Βαΐ συγκεκριμένα γιατί έθιξε το θέμα Ακούω ότι χαιρετίζει τη σύστασή μας να διαφοροποιήσουμε τις υπόλοιπε α, υπόλοιπες με τις απάτες. Εντάξει, ε, φυσικά, γιατί η απάτη είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι απλό διοικητική παρατυπία. Ελπίζω να εγκριθεί η ιδιότητα του Ευρωπαίου Ισαγγελέα γιατί Χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους αυτούς και καλύτερος έλεγχος να μπορούν να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στον πολίτη. Να αρχίσουμε τη συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ομιλητής, η κυρία Γκρέσλε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ συμφωνώ με αυτούς που ε, που λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Θα ήθελα και εγώ να μπορούσα να συμφωνήσω με αυτού που λένε ότι όλα αυτά πήγε πολύ καλά, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Όλαχ, Όλαφ όσον αφορά την ε, αξιοπιστία των στοιχείων. Υπάρχουν στατιστικές ασάφειες για τις διαδικασίες, για το πόσε περιπτώσει έχει αντιμετωπίσει και αυτέ οι ασάφειες μπορεί να θεωρηθεί κανεί ότι είναι αντικείμενο αλλοιώσεων. η Επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε την έκθεση για τον Όλαφ και τις άλλες εκθέσεις για συστημικά προβλήματα και ελλείψεις να τα αντιμετωπίσει. Χρειαζόμαστε να λειτουργεί η καταπολέμηση των διαφθορών. Αλλά εάν δεν έχουμε σωστές στατιστικές, αν δεν έχουμε σωστή λειτουργία των αρποπτικών αρχών, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ε, αποτελεσματική πολιτική. Πρέπει οπωσδήποτε να λάμψει η αλήθεια, αυτό πρέπει να αναφερθεί. Αυτό ισχύει και για την ε, διάσκεψη που έγινε στη χώρα της Επιτρόπου. Είχαν ζητηθεί 605.000 ευρώ και τελικά το κόστος ήταν 136. Νομίζω ότι αυτή η περίεργη αντιμετώπιση των στοιχείων είναι απίστευτη. Αλλά αυτά που κάνετε εσείς ε, κύριε Επίτροπε είναι μια σημαντική αρχή και ελπίζω να δώσετε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι τιμή μου, αλλά είναι και ευχαριστησή μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί είναι πάρα πολύ πλήρης και λογική η έκθεσή του και νομίζω ότι φωτίζει όλες τις γωνίες αυτού του θέματος ε, για την έκθεση για τα συμφέροντα οικονομικά της Ένωσης. Όσον αφορά τη χρήση του 2013, είναι τελευταία χρονιά που αφορά το πολιτή προπολογισμό. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ασόρευση των πληρωμών. Οπότε έχουμε και σχετικά κάποιε αυξήσει σχετικά με το 2012, τα οποία είναι στο φυσιολογικό πλαίσιο. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλούμε για συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα το πολιτέ πλαίσιο θα πρέπει έτσι να το δούμε και να μην κοιτάμε την κάθε χρήση χωριστά και μην κάνουμε σαλαμοποίηση γιατί έτσι παραποιούμε την αλήθεια. Οπότε ευχαριστώ φυσικά τον εισηγητή γιατί εις βάθος εξέτασε το θέμα των εσόδων γιατί τόσα χρόνια κι εμείς προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τις δαπάνες, πώς θα δαπανούμε λογικότερα. Αλλά οπότε έτσι υπάρχει ένα τέτοιο πνεύμα το οποίο το έχει σπαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αλλά και τα κράτη-μέλη και αυτό το οποίο παραβλέπουμε είναι τι γίνεται με τα έσοδα. Τι γίνεται επομένω με τα χρήματα που μπαίνουν στον προπολογισμό, γιατί εδώ πέρα ε, υπάρχουν κάποια σημεία ενισχυτικά δηλαδή για το 2013 όσον αφορά τα τελωνιακά δεν ήμασταν όσο αυστηροί έπρεπε οπότε εδώ πέρα επιδέχονται τα πράγματα βελτίωση λαθρεμπόριο σιγαρέτων εδώ πέρα έχουμε αύξηση συνολική 10 δις ευρώ, όπως είπαμε, και, και γι' αυτό και έχουμε και το πρόγραμμα Juncker για να καλύψει και αυτό. Οπότε ελπίζουμε αυτά να ανακτηθούν παρά, παρά λέγω, αυτό που είπε ο κύριε Γκρέσλερ, ε, ότι η Όλαφ απέσπασε κάποιες πολύ σημαντικές ε, επιτυχίες αυτά τα 68 ε, τα λαθρέα καύσιμα, κατάσχεση φορτίων ε, κοκαίνης. Επομένως, μπράβο στην Όλαφ. Καλά τα πάει. Επίσης, το ε, σύστημα ελέγχου των προϊόντων που επιδέχονται έμεσους φόρους έχει κάποια προβλήματα. Οπότε χρειάζεται τώρα μια καινούργια διαδικασία για να τα βελτιώσουμε. Μια διαπίστωση τώρα που μας τρώει χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή έχουμε τις μη δόλιες παρατυπίες που αυξάνονται και επομένως αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Αλλά αυτό γίνεται πολλές φορές από άγνοια διατάξεων ή από την πολυνομία. Ελπίζουμε επομένως ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να λύσουμε τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω, ελπίζω λέω. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Τσαρνέτσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε κυρίες και κύριοι. Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μάθει για το πώς χρησιμοποιείται το κοινοτικό χρήμα. Τώρα μιλάμε για 2 δις ευρώ. Εκείνα το οποίο έχουν διασπαθιστεί με τρόπο παράτυπο, για να το πω πολύ διπλωματικά. Ε, αυτό δεν θα το αρέσει καθόλου. Και με μεγάλη μου χαρά μαθαίνω ότι δεν πρόκειται εδώ περί δολίων παρατυπιών, περί απατών. Όμως είπαμε την άλλη ότι έχουμε την αύξηση αυτών των παρατυπιών κατά 63%. Πάντως, όπως βλέπουν τα πράγματα οι φορολογούμενοι, αυτές οι λεπτομέρειες είναι αδιάφορες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι τελικά διασπαθίζονται, χάνονται αυτοί οι πόροι. Βεβαίω και έχει καταγάγει πολλές επιτυχίες η Όλαφ και συμφωνώ με όσα είπε η προλαλή σας συνάδελφος. Όμως από την άλλη μεριά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το πώς θα μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε την δραστηριότητα της ε, Όλαφ. Μπράβο της για την καλή συνεργασία με τα κρατη που είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν. Είναι τελικά θέμα πολιτικού βολονταρισμού, πολιτικής βούλης με τα κράτη-μέλη. Ε, από εκεί εξαρτάται το αν καταπολεμείται η, απάτη. Και βέβαια υπάρχει πολυμορφία στο ότι γίνεται από κράτος σε κράτος. Άρα θα πρέπει να πάμε στην πατρίδα μας και να ρωτήσουμε την κυβέρνησή μας τι κάνει, πώς εντοπίζει την απάντηση. Κύριε Ζάνη, θέλετε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γιονάτκη. Τζερνάτκη μάλλον. Ε, δέχεστε κάρτα από τον κύριο Τζάνι, το ανάποδο. Κύριε Τσάρνετκι, αναφέρατε ότι οι αθέμητες πληρωμές μέχρι και 2 δισεκατομμύρια έχουν σημειωθεί αλλά φαντάζομαι ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας. Εσείς ή το πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείτε συμφωνείτε να καθοριστεί η θέση του Ευρωπαίου Ισαγγελέα. κύριε Τσαρνάτσκι. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Πολύ σημαντική ερώτηση σας. Δεν, είμαι, δεν έχω πιστεί πλήρως για τη χρησιμότητα μιας ακόμη υπηρεσίας ή θέσης που θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις δικαιοδοσίες άλλων όπως της Όλαφ. Δεν είναι όμως κακή ιδέα αλλά δεν θα ήθελα να βιαστούμε για να καθορίσουμε αυτή την υπηρεσία τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα πιο αποτελεσματικά τα υπάρχοντα εργαλεία Ωραία. Ο κύριος Τόιρερ δύο λεπτά χωρίς μικρόφωνο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι Καταρχώς, να ευχαριστήσω την Επίτροπο Γεωργίευα για την δραστηριότητά της στον τομέα καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης, οικονομικής διαχείρισης των δαπανών μας. Συμφωνούμε. Και εγώ ως εισηγητής είχα υποβάλει μια έκθεση για ένα προπολογισμό που να βασίζεται στην απόδοση. Πρέπει λοιπόν ο προπολογισμό μας να βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι πολίτες μας περιμένουν οι ενωσιακοί πόροι να δαπανώνται, να δαπανώνται ορθώς. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε και στο μέλλον. Ως ομάδα των φιλελευθέρων απαιτήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς που ήδη έχει. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται οι διακοπές και οι απαιτήσει διορθώσεων ούτως ώστε να απαιτούμε να διορθώνονται οι καταστάσεις. 80% των ενωσιακών πόρων διαχειρίζονται από κοινού μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής και οι διορθώσεις και αναστολές υποχρέωσαν τα κράτη-μέλη να ε, κάνουν καλύτερη διαχείριση και μειώθηκε το ποσοστό λαθών. Όμως υπάρχουν και απάτες με δόλο. Δεν είναι δόλιες όλες οι παρατυπίες, αλλά ορισμένες είναι. Υπάρχουν εγκληματικές προθέσεις και διαδικασίες και αυτές πρέπει να τιμωρηθούν. Ο οργανισμός Όλαφ είναι πολύ σημαντικός, αλλά πρέπει να υπάρχει και σωστός έλεγχός του. Δηλαδή Πρέπει να ενισχυθεί η Εποπτική Επιτροπή. Χρειαζόμαστε επίση και Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τι κατάλληλε προποθέσει. Κράτου δικαίου για αυτόν. Και για την ε, σημαντική καταπολέμηση της φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγής. Αν πάνω από ένα δισεκατομμύριο χάνεται από διαδικασίες ε, φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή, πρέπει να δράσουμε. Γι' αυτό εμεί οι φιλελεύθεροι Ζητήσαμε αυτή την ειδική επιτροπή για τα LuxLeaks και ω κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε η αιχμή του δόρατο τη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Γιατί οι πολίτε αναμένουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτέλου να υπάρξει δράση. Ευχαριστώ. Έχει ζητηθεί μπλε κάρτα για εσά. Τη δέχεστε. Κύριε Τόιρερ, δέχεστε την μπλε κάρτα. Παρακαλώ κύριε. Ο κύριο Έθριτς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύτιμα τα χρήματα των φορολογουμένων και πρέπει να τα φροντίζουμε και να μην γίνονται απάτες. Αλλά δεν θα συμφωνούσατε ότι δεν υπάρχει καμία εντολή κανενός είδους στην Ευρώπη για μια ευρωπαϊκή εισαγγελία το οποίο θα αφαιρούσε εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο που θα μπορούσαμε να το επιβάλλουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία εντολή γι' αυτό. Συμφωνείτε. 30 δευτερόλεπτα κύριε Τόιρα. Η μία, το ένα θέμα είναι ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη Ένωση. Και η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα γι' αυτό. Αλλά το αποφασιστικό θέμα είναι, όπω στη χώρα σα, εάν θα πρέπει να αφαιρεθούν αρμοδιότητε από αυτέ που έχει η Ένωση. Για παράδειγμα, η ιστορική ασφάλεια. Και τι θα μα ωφελούσε αυτό. Το έγκλημα δεν σταματάει στα σύνορα. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία λοιπόν. Και όλα αυτά πρέπει να βασίζονται σε κράτο δικαίου. Οπότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα χρήσιμο όργανο και σας καλώ και στον Ομένο Βασίλειο να προωθήσετε αυτή την ιδέα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επανερχόμεθα στο κατάλογο μιλητών από πλευράς των πολιτικών ομάδων η κυρία Άντερσον από πλευράς Γκούε. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Οι παρατυπίες που σημειώθηκαν το 2013 δεν είναι μικρές. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να τις καταπολεμήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό να προστατέψουμε το, τα συμφέροντα, συμφέροντα της Ένωσης. Και μάλιστα σε εποχή λιτότητας. Δυστυχώς το δημοσιονομικό πλαίσιο 14 με 20 αντιπροσωπεύει μειωμένο προϋπολογισμό, τον πρώτο μειωμένο σε 17 χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν και αυξημένη διοικητική δυνατότητα για να καταπολεμήσουμε τις παρατυπίες. Να μην το αγνοούμε και αυτό. Και χρειάζονται κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Αλλά έχω σοβαρές ανησυχίες ως προς τον ορισμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα το επιχείρημα είναι ότι θα καταπολεμήσουμε έτσι διαμεθοριακά εγκλήματα. Ναι, φυσικά, αλλά θα σημαίνει και αυτό πρόσθετες δαπάνες. και είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει τίποτε παραπάνω από ότι τα κράτη-μέλη σε συνεργασία θα μπορούσε μάλιστα θα έλεγα να υπονομεύσει το σύστημα δικαίου που ισχύει στις Βρετανικές νήσους. Ευχαριστούμε. Για τους πράσινους ο κύριος Γιάβορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Μετά από μια μακρά και δύσκολη συζήτηση, οι πράσινοι αποφάσισαν να στηρίξουν την έκθεση που συμπεριλαμβάνει όμως και τις επικρίσεις μας για την Όλαφ. Ε, δεχόμαστε τη χρήση των προστήμων και κυρώσεων για την καταπολέμηση των ε, παρατυπιών και των, της απάτης και για να υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα αλλά με ελάχιστοποίηση του κινδύνου να αυξηθεί το φορολογικό βάρος των πολιτών. Από τις διαμεθοριακές απάτες που διαπιστώθηκαν το 2013 βλέπουμε ότι χρειάζεται επαρκής νομοθεσία ή διευθέτηση τουλάχιστον και για χώρες όπως την Ουγγαρία τη δική μου η προστασία εκείνων που είναι διατεθειμένοι να παράσχουν πληροφορίες είναι ανεπαρκής στην ε, Ουγγαρία ή τους λεγόμενους whistleblowers και τέλος θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η ύπαρξη, να υπάρξει ένα μια υπηρεσία Ευρωπαίου, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρέπει όμως γι' αυτό να πείσουμε και το Συμβούλιο και τους Ευρωπαίους πολίτες ότι θα ήταν αυτό προς το συμφέρον του φορολογούμενου και όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε Πρόεδρος. Η FTD. Κύριος Βαλίνα Λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επομένω, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την απάτη και σε αυτό συμφωνούμε όλες οι πολιτικές ομάδες. Εγώ όμω, ελκύω την προσοχή σε κάτι άλλο. Τι γίνεται όσον αφορά τη διαχείριση του χρήματος για κάποια προγράμματα τα οποία πρόκειται να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Juncker. Γιατί έχουμε εδώ και τα λόμπι ε, και κάποια άλλα έργα τα οποία αφορούν την αποθήκευση του φυσικού αερίου και άλλα προγράμματα τα οποία γίνονται για το περιβάλλον αλλά πολλές φορές έχουμε κάποιες απώλειες πόρων λόγω κάποιων αισιόδοξων μελετών και αυτά είναι χρήματα τα οποία χάνονται. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις προκαταβολές στους ιδιώτες και θα πρέπει επομένω να υπάρχει διαφάνεια ούτω ώστε να δούμε πώς θα γίνεται η σωστή διαχείριση από τα κράτη-μέλη. Κάθε ευρώ το οποίο ε, ε, ε, το οποίο πρέπει να φέρνει θέσει εργασία και να μην πηγαίνει σε χάρες. Επόμενος. Η πρόκειται περί πηγη απατών εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι. Δεν Και θέλουμε τώρα για την απάτη του ΦΠΑ. Πρόκειται για δεκάδες δι όσον αφορά τη Γαλλία. Πρόκειται για αυτές τις παρατυπίες και τις απάτες που εντοπίζονται και μιλάμε 309 εκατομμύρια και 160 εκατομμύρια που έρχονται από την πολιτική κοινωνική συνοχή. Να, μια ε, αγαστή ε, επενδυτή πολιτική φέρνει απάτη. Και έτσι λοιπόν βοηθάται η κυκλοφορία και το πλήσιμο του χρήματο, χωρίς να υπάρχει κάποιο μεταφορά πόρων σε επίπεδο κρατών μελών. Να, τώρα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά έτσι πρόκειται να αφαιρεθεί κάτι που είναι εθνική κυριαρχία, δηλαδή η δικαιοσύνη. Κανείς δεν πρόκειται να ελέγχει μας το θα γίνει. Ζήτω η Ευρώπη των δημοκρατικών κρατών. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, λέει ο κύριο Στεχόσκη. Η διαφάνεια και η τιμιότητα είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι, σημαίνουν ποιότητα στη ζωή. Το ίδιο σημαντικά όπως η δημοκρατία και η ελευθερία. Άρα θα πρέπει για να είναι αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τιμά αυτές τις αξίες. Απειλούνται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης από τη διαφθορά, τη διάθεση προϊόντων εγκλήματος, τις απάτες και άλλες παρανομίες. Επομένως τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι όχι μόνο να επικρίνουμε την Ένωση ή την Επιτροπή κλπ. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνουν τα ίδια τα κρατημέλη, τα οποία πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αποφασιστικότητα και να κόψει την χρηματοδότηση και τα κονδύλια. Α, έχετε όμως μία περώτηση, θα έχεστε. Α, μάλιστα. Καλά να μας τα είπατε, Λυκείο Σεφερτή για το ότι πάντοτε δεν πιάνουν τόπο τα κοινωτικά χρήματα. Επέστε μας ένα παράδειγμα για κάτι που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα θεωρούσατε ότι θα ήταν πιο σωστή η δαπάνη αν γινόταν σε επίπεδο κρατών μελών. Απάντηση. Αγαπητέ Άρνοντ. Δεν νομίζω ότι για να αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μπορεί να διαθέσει η ίδια τους πόρους. Εάν θέλει να είναι ισχυρή, θα πρέπει να μπορεί να διχειριστεί χρήμα. Απλώς χρειάζεται σωστή πολιτική. Πάντως νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο ρωτάτε. Αλλά μην απευθύνεται σε μένα αυτό το ερώτημα. Εγώ είμαι και θέλω ισχυρή Ευρώπη. Βον, ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και ιδιαίτερα για το ότι υπογράμμισε το θέμα των ε, εσόδων. Πολύ συχνά ασχολούμεθα με τις δαπάνες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα έσοδα. Μόνο ένα 2,9% βέβαια είναι αντικείμενο απάτης, αλλά αυτό είναι 60 εκατομμύρια. Και υπολογίζεται ότι τα κράτη-μέλη χάνουν 10 δις το χρόνο λόγω του λαθρεμπόριου σιγαρέτων μόνο. Και επειδή είναι τόσο χαλεπή η καιρή από οικονομική άποψη, είναι απόλυτα ζωτικό να πάρουμε πίσω ακόμη και το τελευταίο ευρώ για να επενδύσουμε στις θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία με τις ε, βιομηχανίες σιγαρέτων για να καταπολεμήσουμε αυτό το λαθρεμπόριο. Και θα πρέπει να έχουμε και μία μελέτη για το πώς μπορούμε να παρακολουθούμε και να ανοιχνεύουμε τα σιγαρέτα. Όλα αυτά τα μέτρα ελπίζουν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ, πάμε ο μιλητής, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε Γεώργιεβα, στη Σλοβακία η διαφθορά υπάρχει σε, κάθε, σε σχέση με κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ενωσιακά χρήματα. Και αφού είστε κι εσείς από τη Βουλγαρία φαντάζομαι γνωρίζετε τι εννοώ. Οι θύνοντες, οι πολιτικοί, οι πιο γνωστοί πολιτικοί εμπλέκονται σε τέτοια σκάνδαλα. Επομένως δεν γίνονται επαρκείς έρευνες. Τον περασμένο χρόνο υπέβαλα μόνος μου 13 αιτήματα έρευνας από την Γιάννολαφ. Αν είστε σοβαροί ότι θέλετε να καταπολεμήσουμε την απάτη, τότε καταργήστε αυτά τα άχρηστα ποσά. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες τους δίνουν συνεχώς λεφτά. Δεν είναι αυτό ο τρόπος, δεν είναι σοσιαλιστικό το η σοσιαλιστική λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, το θέμα θα συζητιέται επί πολλά χρόνια γιατί παραμένει αλήθεια ότι με ευρωπαϊκά χρήματα στα χρήση των ευρωπαϊκών χρημάτων σημειώνονται και απάτες και η Κομισιόν δεν έχει λιγότερες περιπτώσεις κάθε χρόνο αλλά όλο και περισσότερες. Γιατί αυξάνεται μεν η υποστήριξη προς την Ένωση αλλά αυξάνεται και η γνώση των εγκληματιών για το πώς να απατήσουν ε, την Ένωση αποτελεσματικότερα. Πρέπει λοιπόν να νομοθετήσουμε λογικά για να βοηθήσουμε στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που διαθέτουμε. Δεν πρέπει νομίζω να έχουμε αυταπάτες ότι ε, μαγικά θα λυθεί το πρόβλημα της διαφθοράς αλλά πρέπει να ζυγιάσουμε τα πράγματα ακριβώς και το σωστότερο θα ήταν να υπάρχει να δημιουργηθεί μια θέση εισαγγελέως αλλά με περιορισμένες δικαιοδοσίες ο κύριος Άγνοτ η έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης είναι τρομερή βλέπουμε τον, ότι ο αριθμός των απατών έχει αυξηθεί. Μιλάμε για 1609 απάτες. Και αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε, ούτε να το κρύψουμε. Δεν έχουμε κριτήρια σαφή. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει κατασπατάληση χρημάτων και να μην το ξέρουμε. Τι θα σήμαινε όμως αποτελεσματική αντιμετώπιση πρόληψη. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι η φύση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι τόσο μακριά από τον πολίτη ώστε γίνονται τόσο, γίνεται τόσο δύσκολη η αναγνώριση καν του προβλήματος, πόσο μάλλον η λύση. Η λύση λοιπόν είναι να υπάρχει πραγματική λογοδοσία. Ο κύριος Ζάλκ. Για ένα λεπτό. Δεν απουσιάζει. Κύριος Σαρβαμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έκανε καλή δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάθεση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα για την Όλαφ. Ο της είναι η πρόληψη της απάτης και όμως επιδέχεται βελτίωση ο τρόπος λειτουργίας της. Εμείς έχουμε επικρίνει την Όλαφ, αλλά βέβαια θα πρέπει να ε, συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί την Όλαφ ε, ανεξάρτητο, ανεξάρτητη υπηρεσία. Επομένως χρειάζεται αξιοπιστία σε σχέση με τις ε, πληροφορίες για το τι κάνει η Όλαφ και επομένως οι έρευνες της Όλαφ να είναι πιο αποτελεσματικές. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πάντως ε, πολλές φορές ε, κλείνουν τα μάτια σε τέτοια προβλήματα και είδαμε τι έγινε. Έχουμε τις τροπολογίες που υπέβαλαν 12, 13 και 14 τις υπέβαλαν εκ νέου. Αυτό δεν βοηθάει ούτε την Όλαφ, ούτε την πρόληψη της ΑΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λόγια τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να επιδείξει σκληρή στάση κατόπιν αυτών που είπε η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Το να περικοπούν οι καταβολές στα κράτη-μέλη είναι σκληρό, αλλά θα πρέπει να δούμε με τη μέτρα, μπορούμε να έχουμε σωστή χρήση των πόρων της Ένωσης. Ευχαριστούμε. Και τον έλεγε κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που προετοίμασαν την έκθεση αυτή. Το... Πριν από μερικά χρόνια είχα και εγώ συγγράψει μια ανάλογη έκθεση και γι' αυτό γνωρίζω καλά το θέμα το 11. Η Ένωση είχε χάσει τότε στην έκθεσή μου τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια και επεστράφησε, επεστράφει μόνο το 24 τις 100 των χρημάτων που αφορούσαν παρατυπίες ή και απάτες. Επομένως πρέπει να υπάρχει περισσότερος και καλύτερος έλεγχος και καλύτερη χρήση των χρημάτων της Ένωσης να υπάρχουν δηλαδή τα σωστά συστήματα στα κράτη-μέλη. Συνεχώς σημειώνεται το πρόβλημα ότι τα κράτη-μέλη δεν χορηγούν πλήρες πληροφορίες. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις που γίνονται, ούτε εφαρμόζονται ομοιόμορφες κυρώσεις και πρόστιμα. Πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Η καταπολέμηση της απάτης είναι το θεμέλιο μιας σωστά δομημένης κοινωνίας. Πρέπει όμως να δεχτούμε το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ είναι υποχρεωμένη εδώ να αναγνωρίσει ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Δεν έχει υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ των εσόδων και της ε, υπερβολικής φορολόγησης των πολιτών σε ορισμένα κράτη-μέλη. Πράγμα το οποίο όθησε σε περισσότερο ασταθείς προϋπολογισμούς. Τα ποσά που χορηγούν στον προϋπολογισμό η πολιτική με κριτήρια αδιαφανή πολλές φορές δεν διευκολύνουν τον έλεγχο αλλά τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος ένα λεπτό. ορίζω την έκθεση αυτή του κυρίου Πυρίνσκι και τονίζω ότι η απάτη δεν είναι πρόβλημα μόνο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απάτη σημειώνονται σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Το υψηλό επίπεδο κατάχρηση δημοσίων πόρων έχει τεχνική φύση. Έχει υπάρξει παραμέληση της ε, σωστής τελέχωσης και κατάρτισης των δημοσίων αρχών και του σωστού εξοπλισμού των. Ναι, μεν ανεβαίνουν οι αριθμοί, αλλά ως ποσοστά έχουν μειωθεί οι παρατυπίες. Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση ωστόσο και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ε, περιπτώσεων απατών. Πρέπει να παραμείνει η πολιτική συνοχή αξιόπιστη και αποτελεσματική μέσω αυτής της αντιμετώπισης. Η κυρία Νταμάτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η έκθεση του κυρίου Πυρίνσκη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λίγα αυτέ τι σκέψει. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δούμε ότι για πρώτη φορά η πολιτική τη συνοχή είναι ο δεύτερο τομέα σε σχέση με τι δαπάνε των προπολογισμών. Αλλά εκεί βλέπουμε ότι όλε αυτέ τι περιπτώσει ε, απάτης μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. 321 τέτοιες δόλειες περιπτώσεις είχαμε, 4.600 μη δόλειες, οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενισχυτικά και θα πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να μειωθούν οι οικονομικές, εδαφικές, κοινωνικές ε, ανισότητες. Η Ιταλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία ε, είναι επικεφαλής του καταλόγου για αυτές τις ε, απάτες και στην Ιταλία έχουμε 72 τέτοιες περιπτώσεις απόπειρας απάτες ή απάτες. Μόνο το 2013 και μόνο για την πολιτική συνοχή. Βέβαια, είναι θετικό το ότι το ανακάλυψαν οι αρχές. Ε, οπότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και όσον αφορά την ε, διαφθορά από τους απάτες αλλά επίση και για, τα, για το, σύστημα της, ε, το σύστημα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Κόβει το μικρόφωνο η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Όμως υπάρχει μία επερώτηση για σας. Δέχεστε, ναι λέει η κυρία Νταμάτο, από τον κύριο Γιάκοβσιτς. Κυρία Νταμάτο, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Έχουμε συνεργαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και έχω να σας απευθύνω την εξή ερώτηση. Σοβαρά έγινε συζήτηση σε σχέση με το πώς θα απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και και να δούμε τι γίνεται με όλες αυτές τις ε, κοινοποιηθεί σε περιπτώσει απάτης που πολλές φορές γίνονται κατά λάθο. Εσείς συμφωνείτε πρέπει να διορθώσουμε τη διαδικασία. Αυτό είναι γεγονός. Και στην Ιταλία, στις περιφέρειες στι λιγότερο αναπτυγμένε, έχουμε ακόμα περιπτώσει τέτοιες απάτη. Τα λειτουργικά προγράμματα μπλοκάρονται και επομένω εκεί χρειάζονται περισσότερο να πάνε σχετικοί πόροι. Να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν οι αρχές και ασχοληθήκαμε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και είπαμε θα πρέπει να πώς γίνεται η πιστοποίηση οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί ελέγχους καλύτερα. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και τώρα το λόγο κυρία Κινέτσι. Έχετε μόνο ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την κυρία Επίτροπο αλλά και τον εισηγητή για το έργο του, για αυτή την έκθεση που τώρα συζητούμε. Και οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για αυτά με αυτά τα εγκλήματα. Τα είδαμε και στην Επιτροπή Κόντ, είδαμε και τις τροπολογίες, ότι η προστασία των συμφωνών της Ένωσης θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για τις πολιτικές της Ένωσης. Είδαμε το πόσο απογοτεύουν αυτά τα αποτελέσματα. Ε, πάει καλύτερα η Όλαφα, αλλά έχουμε ε, έρευνε όλο και περισσότερες και λένε και λιγότερο υπάρχει χρόνο για να γίνουν σχετικέ συστάσει. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ποσοστά τη ε, ανάκτηση. Ακόμα επειδή έχονται βελτίωση αυτέ οι επιδόσει και άρα θα πρέπει να δούμε πώ ε, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ε, χρειάζεται ταχύτητες αποφάσεων, ανεξαρτησία, αμεροληψία. Οπότε έτσι θα πρέπει να φροντίσει την προστασία των συμφερόντων της Ένωση που είναι τελικά χρήματα των φορολογουμένων. Η πρόεδρο. Κύριε Κινέτσο, υπάρχει μια επερώτηση για σας. Τον κύριο Κόβιν Μίκη. Έχετε μισό λεπτό κύριε συζητούμε την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Δεν συζητούμε για την διαφθορά. Δεν θεωρείται ότι χάνουμε πολύ περισσότερους πόρους όσον αφορά τα διοικητικά και τα νομικά, γιατί για τη γνώμη μου 95% των χρημάτων διασπαθίζονται. Και όλες αυτές οι ιδέες και αυτά τα προγράμματα είναι επιβλαβή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κύριε Κινέτσο, για να απαντήσει. Να σας απαντήσω πάρα πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε να φροντίζουμε τα οικονομικά συμφέροντα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη διαφθορά. Χρειάζονται, και οι ενέργειες για το πόνο της και η προστασία των συμφέροντων. Ένα λεπτό κύριο Βοητσεσχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Όλους μας ανησυχεί και με όλους μας ενδιαφέρει το θέμα της ε, υπεράσπισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά γιατί τίθεται ένα θέμα ακαιρεότητα στην καθημερινή ζωή. Χρειάζεται λοιπόν σαφήνεια αυτή είναι η έννοια κλειδί. Οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις υπάρχουν από την Ένωση πρέπει να γίνονται και να δαπανώνται τα ποσά με διαφανή τρόπο και να ξέρουμε τι ακριβώς χρηματοδοτούν ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δυστυχώς η κατάσταση στην πράξη δεν είναι αυτή η θεωρητική που περιέγραψα. Προσπαθώ να βρω, προσπάθησα συγκεκριμένα, να βρω πώς δαπανήθηκαν ε, κάποια ποσά για κάποια θέματα στην Πολωνία και ελπίζω και στο μέλλον να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσουμε την διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάτσεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ένωση ανεπιτυχώς προσπαθεί χρόνια να αντιμετωπίσει τις απάτες. Νομίζω ότι ε, τα τελευταία 20 χρόνια οι λογιστές δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν με τους ε, λογαριασμούς της Ένωσης. Σε οποιοδήποτε ιδιωτικό οργανισμό αυτό θα είχε οδηγήσει στο κλείσιμο. Θα είχε παρέμβει ο εισαγγελέας. Το Ταμείο Συνοχής και η κοινή γεωρική πολιτική είναι οι κύριοι τομείς απατών και οι χώρες με τις περισσότερες παρατυπίες είναι η Ιταλία, η Ρωμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Δανία και η Ελλάδα. Δεν μας εκπλήσουν αυτά τα ονόματα. Εάν δώσουμε τόσα τεράστια ποσά σε χώρες που είναι θεσμοθετημένα ε, διεφθαρμένες, τότε θα βρεθούν εγκληματίες για να αποφεληθούν. Και οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι μου στο Λονδίνο φυσικά ε, σοκάρονται από το πόσο άσχημα δαπανώνται τα χρήματά τους. Και πιστεύω ότι ψηφίζοντας στις 7 Μαΐου UKIP θα βοηθήσουν να βγει η χώρα μου από την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβάν απουσιάζει. Ο κύριος Μπάρεκοφ λοιπόν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Γεωργίευα. Ήχμουν στη χώρα μου πολύ στενά συνδεδεμένος στη δουλειά μου με υποθέσεις κατεπολέμησης απατών και ξέρω ότι μέχρι τώρα όλες οι χώρες που γνώρισα είχαν υποβάλει πληροφορίες για γνωστοποίηση απατών αλλά δεν είχε αντιμετωπιστεί τίποτα. Πρέπει λοιπόν ο μελλοντικό εισαγγελέα να γνωρίζει ότι η υπηρεσία του μπορεί να μην καταφέρει να καταπολεμήσει το έγκλημα. Άρα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται εγκληματική δραστηριότητα. Πρέπει τουλάχιστον να επιτευχθεί να σημειωθούν λιγότερες περιπτώσεις δαπανών. Ένα λεπτό κύριος Μάχ. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας ε, μας δίνει πολλά στοιχεία για τις απάτες, για την κακοδιαχείριση ενωσιακών πόρων. Αυτά είναι χρήματα των φορολογουμένων, ξέρετε. Άρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Φοβάμαι όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο αρνείται να δει το αίτιο που είναι η ο θανάσιμος εφησυχασμός και η βαθιά πίστη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μηχανισμός αναδιανομής πιστώσεων. Γιατί να μην κάνουν την πολιτική για τα θέματα αυτά τα κράτη-μέλη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, για να πληρώσουν για δρόμους, επιτόπου. Γιατί να μην ε, αποφασίσουν οι ίδιοι πολίτες του κάθε κράτους μέλους. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να καταργήσουμε τα ταμεία και να καταργήσουμε τη διαφθορά που επιφέρουν. Ευχαριστώ πολύ να απειλήσουμε στη διαδικασία προσέλκυσης ε, προσοχής του Προέδρου. 13 έχουν στήσει το λόγο, οπότε 8 θα μπορούσε να τον πάρουν, ένα λεπτό θα έχει η κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σωστή δαπάνηση από τον προϋπολογισμό πρέπει να είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εάν ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της Ένωσης. Σωστά δαπανημένα δημόσια χρήματα είναι καλύτερος τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς την Ένωση από ότι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλος. Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία όμως και δεν επιτρέπει αυτό τη σωστή αντιμετώπιση των παρατυπιών. Το ανησυχητικό είναι ο δείκτης που αυξήθηκε το 2013 και που δείχνει ότι η απάτη δεν έχει αποτελεσματικής καταπολέμησης. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και από πού προέρχονται οι απάτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταπολέμηση της απάτης είναι μια προτεραιότητα όσον αφορά την κοινότητα αλλά και τα κρατη Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο μας ενισχύει πάρα πολύ. Πρώτα για μια ήττα κοινωνική και ηθική για το ότι έχουμε κατά διάφορους τρόπους παραβίαση των κανόνων. Και αυτό βλέπουμε ότι υπονομεύει την Ευρώπη. Επομένως χρειάζεται να δούμε πώς θα έχουμε ενιαίο μέτωπο ούτως ώστε να πάρουμε κάποια μέτρα εναρμονισμένα όσον αφορά τις σχετικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Επίσης πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών. Και επίσης όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική οικονομία. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζονται καλύτερες ε, διαδικασίες για να μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται και να κατοπολεμήσουμε τις παρατυπίες. Κύριε Μαριά, έχετε ένα λεπτό. Για των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και το κτύπημα της απάτης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δράση ιδίω σε αυτή τη φάση της έντονης οικονομικής κρίσης. Οι απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και σε ορισμένες χώρες συνδυάζονται με τη δράση της μαφίας του κεφαλαίου, της μάφια καπιτάλε όπως λένε στην Ιταλία έτσι το λαθρεμπόριο καυσίμων το λαθρεμπόριο τσιγάρων οι απάτες σε σχέση με το ΦΠΑ και η φοροδιαφυγή τύπου leaks είναι στην ημερήσια διάταξη. βεβαίως υπάρχουν και οι παρατυπίες που συμβαίνουν όχι από δόλο αλλά καθαρά από αμέλεια. εδώ πρέπει να εντείνουμε την προληπτική μας δράση προκειμένου να αξιοποιήσουμε ορθά τα περιορισμένα κονδύλια των ευρωπαϊκών ταμείων. το γεγονός ότι οι απάτες και παρατυπίες κοστολογούνται στο ύψο των δύο των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το ευρώ του προβλήματος που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε γιατί οι ευρωπαίοι πολίτες δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλε απάτες και παρατυπίες στη διαχείριση των κονδυλίων της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. λεπτό. Δεν έχω καμία πρόθεση να μειώσω τη σημασία της συζήτηση αυτής. Και τονίζω ότι συζητάμε ένα θέμα που αφορά δύο δις σε απάτες και άλλες παρατυπίες. Αλλά θέλω να τονίσω ότι χρειάζονται αυστηρότατες κυρώσεις για όλες τις εγκληματικές ενέργειες και είμαι υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γιατί το έγκλημα είναι διεθνές. Αλλά επίσης ως κάποιος που έχει εργαστεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για πολλά χρόνια, κυρία Επίτροπε, πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Υπάρχουν ε, παράλογες καταστάσεις όπου ε, κάτι θεωρείται απάτη, ενώ ε, στην πραγματικότητα μπορεί να αγόρασαν ας πούμε ξύλινες πόρτες και όχι μεταλλικές, ενώ η προδιαγραφή έλεγε το άλλο και άρα το, συμβούλιο, το συμβόλιο θεωρείται ότι παραβίασε τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιέγας, ένα λεπτό. Βεβαίως πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απάτες και οποιασδήποτε παρατυπίες. Το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί την καλή χρήση των πόρων είναι σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα για να ε, προφυλάξουμε τους ίδιους πόρους μας. Γιατί διαπιστώνουμε όλο και περισσότερες παρατυπίες σε διάφορα ταμεία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε και τον κυτρινισμό ορισμένων. Αλλά ε, διαπιστώσαμε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν πρόκειται για απάτες, αλλά απλώς για παρατυπίες. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι διαδικασίε για την αίτηση πόρων είναι πολύ περίπλοκε. Είναι σαφέ ότι υπάρχουν βέβαια και κάποιε απάτε, αλλά σε ορισμένε άλλε περιπτώσει απλώ ο καθένα δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ ζητάει. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν και τι διαδικασίε και του ελέγχου. Κάτι άλλο είναι πώς αξιοποιούμε τους ίδιους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και πολλές χώρες, έχει οργανωτικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλά ε, ε, σχήματα για να αποφεύγουν διάφοροι να πληρώνουν φόρους. Η κυρία Μόη. Εγώ θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο πρόβλημα το πώς θα πανώνται κάποιοι πόροι που απευθύνονται σε κράτη-μέλη και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Εγώ προέρχομαι από ένα νησί, την Σαρδίνια, που είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά το λάθος για την κοινοποίηση των πόρων από τα κοινωνικά ταμεία. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τις άλλες περιφέρειες και καλύπτονται έτσι ε, πάρα πολλές λαθροχειρίες ε, ότι είναι δήθεν ε, στα περιθώρια, στα προστασία της ζωής. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα έχουμε μέσω της ε, τοπικής διεφθαρμένης πολιτικής διασπάσεις των πόρων. Είναι δύσκολο το έργο της όλων αλλά η κατάσταση είναι πια αφόρητη και θα πρέπει να γίνει για λάση αυτή η κατάσταση για πάτε και για διαφθορά όσον αφορά τον ευρωπαϊκό κορβάνα. Οπότε θα πρέπει να προσέχει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πιο αποφασιστική και καλύτερα από ό,τι κάνει τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέιλε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι σκανδαλώδες το ποσό, το χρηματικό το οποίο χάνεται. Χάνεται λόγω των διαφορετικών παραλλαγών απάτης που συμβαίνουν. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα και όπως είπε και ε, ο εισηγητής χάνουμε δύο δις ετησίες λόγω των απατών, των παρατυπιών κλπ. Και είναι σαφές ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές. Έτσι ίσως καταπολεμήσουμε καλύτερα την απάτη. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί μια πιο σωστή νοοτροπία και καλύτερη νομοθετική πλαισίωση των προγραμμάτων. Ίσως έτσι οι παρατυπίες και οι απάντες μειωθούν. Η Πρόεδρος. Ένα λεπτό κυρία Πησιάνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δίνει ε, ένα πλαίσιο θετικό για την κατάσταση αυτή της απάτης όσον αφορά το ότι έχουν αυξηθεί οι παρατυπίες αλλά έχουν, ε, έχουν σχετικά πόσα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά το το 2013 Είχαμε 69 τέτοιε παρατυπίες, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σημαντικέ ε, στην ε, Γεωργία αλλά και στην Αλία. Και εγώ εδώ θέλω να σας ξαναπώ ότι δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε ούτε ενό ευρώ διασπάθηση από τους κοινοτικού πόρους με τέτοιου είδους συμπεριφορές ε, παράνομες και παράτυπες. Άρα θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη θα πρέπει στη ρίζα να χτυπήσουμε το κακό αυτών των συμπεριφορών, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή σωστών πρακτικών για να δούμε ε, με την Όλαφ πώς θα συνεργαστούμε ε, με την Όλαφ ε, και θα πρέπει και τα άλλα κρατημέλη να συνεργαστούν οπότε θα πρέπει να υπάρχει καταστολή τιμωρία και να βοηθήσει και με ποινικέ διατάξεις και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόεδρος. Έχετε μία επερώτηση, κυρία. Αποδέχεστε. Τον κύριο Βάλιο. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να ρωτήσω την συνάδελφο του. Γνωρίζει ότι οι έλεγχοι για τα τα ταμεία γίνονται από τις εθνικές αρχές και θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιου ελεγχού, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι για να γίνουν στι περιφέρειε αυτή η ελέγχη. Και εδώ και πολλά χρόνια έτσι έκαναν οι περισσότερε κυβερνήσει στην Ιταλία. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει ούτω ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να ξέρουν οι πολίτε πώ γίνεται η διαχείριση των πόρων. Μισό λεπτό για να απαντήσετε κυρία. Ευχαριστώ κύριε Βάλη για την ερώτηση. Οπότε τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας τονίσω το ότι σας έχει διαφύγει πως εμείς όσον αφορά την πολιτική καταπολέμηση απάτης είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Από το 2007 υπάρχει συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων και έτσι κυνηγάμε την απάτη. Βεβαίως και όλα αυτά επιτέχονται βελτίωση και δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ε, πραγματικότητα γιατί ακόμα έχουμε πολλές περιπτώσεις απάτες. Αλλά γίνονται βήματα πρόοδου και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα έτσι κλείνει η διαδικασία ΓΕΣΔΙ και τώρα έχει το λόγο επίτροπος και Γεωργίευα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για όλα τα σχόλια που έγιναν. Έχουμε την τεράστια ευθύνη και υποχρέωση προς τους πολίτες μας να χρησιμοποιούμε τα χρήματα με τρόπο σωστό και χωρίς καμία κατασπατάληση. Α, στην πραγματικότητα ο αριθμός απατών για τις δαπάνες έχει μειωθεί λιγάκι από το 0,90 της 100 στο 0, ε, μάλλον, στο 0,20 έχει αυξηθεί μάλλον λιγάκι. Αλλά και αυτό το λίγο είναι υπερβολικό. Ακούστηκε το σχόλιο ότι ότι δεν υπογράφονται οι λογαριασμοί μας. Υπογράφονται κάθε χρόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Ακόμη όμως υπάρχουν πολλά λάθη. 4,7% είναι υπερβολικά ψηλό ποσοστό γιατί είχαμε θέσει, στο δικαστήριο είχε θέσει ως ανεκτό όριο το 2%. Πρέπει λοιπόν είπε επίσης στο δικαστήριο να απλοποιηθούν οι κανόνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο έτσι θα μειωθούν τα λάθη ή μάλλον δεν είναι ο μόνος λόγος η απλοποίηση για να μειωθούν τα λάθη αλλά και για να υπάρξει καλύτερη χρήση των χρημάτων. Όταν τα πράγματα είναι πολύπλοκα είναι πιο εύκολο να γίνουν απάτες. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι για αυτόν τον λόγο προσβλέπουμε στο Κοινοβούλιο ως εταίρο για να μας βοηθήσει σε αυτή την απλοποίηση. Δυστυχώς αρχίσαμε από απλούστερους κανόνες και να καταλήξουμε σε πιο πολύπλοκους. Αλλά και μέσα στα πλαίσια του Πολδίπ νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με την απλούστευση καλύτερα τα χρήματα που διαθέτουμε. Συμφωνώ απόλυτα με εκείνους που είπαν ότι είναι σημαντικό να δούμε και την πλευρά των εσόδων διότι εκεί η τάση που σημειώνεται είναι η αντίθετη. Έχει αυξηθεί η, λιγάκι η απάτη εκεί. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας γιατί είναι χρήματα που προέρχονται από τις χώρες μέλη και είναι ποινικό αδίκημα. Ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, συμφωνώ. Αλλά η πρόληψη της, του λάθους είναι κάτι φυσικά καλύτερο από το να χρειάζεται κανείς να το διορθώσει αλλά υπάρχουν και οι απάτες και ισχύει αυτό και για τις απάτες. Η θέση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα νομίζω ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και θέματα απάτης για το ΦΠΑ και έτσι θα είμαστε πιο πολύ και όχι λιγότερο αποτελεσματικοί γιατί το είπαν και αυτό μερικοί γιατί θα μπορούσαμε έτσι να προστατεύουμε καλύτερα τα συμφέροντα της Ένωσης και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα είναι τα συμφέροντα των φορολογουμένων γι' αυτό όμως πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι γι' αυτό ζητήσαμε η Επιτροπή Εποπτείας να εξετάσει και το θέμα της αξιοπιστίας των δεδομένων που διαθέτουμε που μας χορηγούν όλες οι άλλες υπηρεσίες. Να μην ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Εμένα με ενδιαφέρει βέβαια τελικά το αποτέλεσμα. Η συζήτηση αυτή φυσικά θα συνεχιστεί. Δεν θα σταματήσει ποτέ η δράση μας και τελικά θα κριθούμε από τα έργα και όχι από τα λόγια μας. Ευχαριστούμε. Και τελευταίος ο εισηγητής κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτής της προσπάθειας που κάνουμε είναι να καταλήξουμε στην ε, λειτουργική και αποτελεσματική συνεργασία Κοινοβουλίου και Επιτροπής για να αντιμετωπίσουμε όντως τις παρατυπίες, τις απάτες, γιατί είμαι πεπισμένος ότι η Επιτροπή μέσω της κυρίας ε, Γεωργίευα έδωσε μια σαφή υπόσχεση ότι δεσμεύεται να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους. Άρα πρέπει να τη στηρίξουμε πλήρως. Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε που λέει ότι πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα των στατιστικών μας και καλό τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη τα στοιχεία. Από το 1,7 δις των δαπανών που είναι αντικείμενο παρατεπιών είναι το 1,34% των συνολικών δαπάνων. Δηλαδή αυτό το 1,7 είναι το 1,34. Δηλαδή 98,1% των δαπανών μας εκταμιεύθησαν ε, νομοτύπως. Για τους ίδιους πόρους. Ανακτήσαμε 380 εκατομμύρια. Μα τα λέει η έκθεση. Μην ανησυχείτε, τα λέει η έκθεση. 380 εκατομμύρια ήταν αντικείμενο παρατυπιών. Ήταν 1,6% των παραδοσιακών ίδιων πόρων. 1,86, συγγνώμη. Επιπλέον το 2013, ο όγκος των παρατυπιών που διεπράχθησαν μειώθηκε κατά 30% σε σχέση με το 12. Και των δαπανών, το ύψος των, δαπαν, των, ε, των απατών κατά 30%. Ναι, μεν αυξήθηκε ο αριθμός παρατυπιών, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προβούμε σε περισσότερες ενέργειες και, και έρευνες, αλλά τώρα να αυτομαστιγωνόμαστε δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστούμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε. Λίγη εδώ και αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. αύριο. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Διεθνή Διάσκεψη για τον ιό του έμπολα της 3ης Μαρτίου 2015. Κυρία Κανίνια Λουκασένκα.